Ε, ολοκληρώθηκε η συζήτηση και αυτή η ψηφοφορία αύριο στις 6 ώρα. Κυρίες και κύριοι, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, έκθεση Μπαχ. Νομίζω πως είναι το αποκορύφημα της βραδιάς, αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κινητικότητα είναι πυλώνας της σύγχρονης κοινωνίας, κάτι το οποίο ε, φαίνεται καθώς τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση ε, των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Ήδη η Κομισιόν πριν από 10 χρόνια έχει τονίσει την ανάγκη ενιαίων δικαιωμάτων των επιβατών. Εν τω μεταξύ έχουμε έξι κανονισμούς για το θέμα αυτό, όμως οι εμπειρίες των τελευταίων ετών δείχνουν πως οι υφιστάμενοι κανονισμοί αφήνουν παραθυράκια και ασάφειες, κάτι το οποίο οδηγεί σε μια μη ενιαία εφαρμογή από τις ε, επιχειρήσεις ε, και τα δικαστήρια. Οπότε χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Κομισιόν να προσαρμόσει όλες αυτές τις ε, διατάξεις, να ενισχύσει την εθνική τους εφαρμογή και να δώσει περισσότερες πληροφορίες στους επιβάτες για τα δικαιώματά τους. Αυτή τη στιγμή ένας ενιαίος κανονισμός δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχει αρκετή εμπειρία για τους επιβάτες πλοίων και λεωφορείων. Μεσοπρόθεσμα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθήσουμε για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Οπότε ζητάμε να ισχύουν τα ίδια δικαιώματα και για τους ε, τέσσερις ε, τρόπους και μέσα μεταφοράς χωρίς βεβαίως να παραβλέπουμε τις ιδιαιτερότητες τους και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα και την θέση της κάθε εταιρεία η οποία εκτελεί μεταφορές. Οπότε θα πρέπει και η Κομισιό να επεξεργαστεί κάποιες κατευθύνριε γραμμές έτσι ώστε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την εκπλήρωση της σύμβασης μεταφοράς, την πληροφόρηση, την άμεση βοήθεια και βεβαίως οπωσδήποτε το να μην εξασθενήσουν τα εφιστάμενα δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια σημεία της έκθεσης. Όσον αφορά την πληροφόρηση και την διαφάνεια λέγεται πως θα πρέπει να είναι άμεση και ξεκαθαρή πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης να εκπαιδευτεί το προσωπικό το οποίο στελεχώνει τα σημεία πληροφοριών. Θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Όσον αφορά δε τη χρήση και εφαρμογή των αυτών των δικαιωμάτων, σημασία έχει και η συμπεριφορά των εθνικών αρχών. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει, θεωρώ εγώ, μια ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για να υπάρξει πιο αποτελεσματική εργασία εδώ. Θα μπορούσε να υπάρχει μια κεντρική ηλεκτρονική υπηρεσία παραπώνων. Επίσης ε, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την αστική ευθύνη και την ε, χρήση του όρου έκτακτες συνθήκες. Εδώ πέρα νομίζω πως πρέπει να συμμορφωθούμε με την ομολογία του ΔΕΚ. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ε, των ανθρώπων με αναπηρίες και περιορισμένη κινητικότητα ειδικά όσον αφορά τα ταξίδια με παραπάνω από ένα μέσα μεταφορά. Τέλος, με την οικονομική κρίση είχαμε αύξηση των χρεοκοπιών αεροπορικών εταιριών και εδώ πέρα επιτέλους θέλουμε συγκεκριμένες προτάσεις από πλευρά Κομισιόν. τέλο. θα ήθελα να αφαιρθώ στην αύξηση των διατροπικών ταξιδιών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν δικαιώματα διασύνδεσης για όλα τα μέσα μεταφοράς και τις εταιρείες. Βεβαίως, προϋπόθεση είναι να λειτουργούν καλά οι διατροπικές αυτές ενθέσεις. Τέλος, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις ε, συνεισφορές τους, με στήριξαν και ε, με βοήθησαν να αποκτήσει ουσία αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε στη διαδικασία KHDI. Κυρία Μπασέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω κυρίως να χαιρετήσω την ε, ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών. Πρέπει η εφαρμογή τους να είναι προτεραιότητα, να γίνεται εξαντλητικά και ομοιόμορφα για να μην υπάρχουν συγχύσεις. Οι ταξιδιώτες έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται μονίμως για τα δικαιώματά τους. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς, απλές και προσβάσιμες. Πρέπει επίσης να αυξηθεί η διαφάνεια σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται για να σταματήσουν οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Υπογραμμίζω ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να έχουν υψηλό επίπεδο προστασίας και οι εθνικές αρχές ελέγχου πρέπει να παίξουν το ρόλο που τους ανατίθεται. Η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα ε, επιβατών όλων των μέσων μεταφοράς θα επιτρέψει καλύτερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς είναι ε, πολύ επίκαιρο. Υπάρχει το θέμα των ε, ενημέρωσης, τα δικαιώματα των ε, ατόμων με περιορισμένη ε, κινητικότητα ή με προβλήματα κινητικότητα. Και βεβαίω δεν αναφέρεται ούτε μία φορά το θέμα των δημοσίων υπηρεσιών. Το πρώτο και βασικότερο δικαίωμα των επιβατών και όλων των ανθρώπων είναι το δικαίωμα σε ένα υψηλή ποιότητα σύστημα μεταφορών ε, που να είναι αποτελεσματικό, σύγχρονο και σε ε, καλή τιμή. Αυτό σε χώρε όπω το δικό μου έχει υπέρθει καταστροφή των δημοσίων συστημάτων μεταφορών που έχει προ... Προ... οφείλεται στην ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνέ Σωματικό Ταμείο έχει οδηγήσει σε κατάργηση υπηρεσιών, ε, αύξηση τιμών, ε, ε, απολύσεις και τελικά θα μειωθεί η παροχή υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δικαιώματα επιβατών αν δεν μιλήσουμε για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Φερέρα. Κύριος Πάνκη για ένα λεπτό. Θα ήθελα να συγχαρώ κυρίως τον συνάδελφο Μπαχ διότι, ε, που ήταν ο εισηγητής γιατί πέρα από το γεγονός ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τη διαφάνεια των ε, ε, της πληροφόρησης των επιβατών θα πρέπει να κοιτάξουμε να εναρμονίσουμε και τις εθνικές νομοθεσίες. Είναι αξιέπαινο η προσπάθεια του να έχουμε μία τράπεζα δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των εθνικών τραπεζών δεδομένων. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ο τουρισμός. Πράγματι θα πρέπει να παρέχουμε όλο ένα και μεγαλύτερες υπηρεσίες ε, ποιότητας και πρέπει να εγγυωμηθούμε και έναν ε, αηφόρο τουρισμό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν οι ταξιδιώτες δικαιώματα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ευχαριστώ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κυρία Τσίκαου. Ευχαριστώ. Να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε τους κανόνες για τα δικαιώματα των πολιτών στις μεταφορές και θα συνεχιστεί μέχρι το 2014 αυτή η πληροφορική, πληροφορική εκστρατεία πληροφόρησης προς τους ε, Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν. Θεωρώ ότι η καμπάνια αυτή, αυτή η εξαρτία θα πρέπει να επεκταθεί και στους αναπήρους διαφημίζοντας δηλαδή τις, ε, τα δικαιώματα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους και θέτοντας, ε, ε, δημιουργώντας επίσης σημεία πληροφόρησης μέσα στα αεροδρόμια που θα δίνουν πληροφορίες για τους ανάπηρους. Υπάρχει επίσης πρόβλημα μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχουν οι αεροπορικές εταιρείες. Θα θέλαμε να υπάρχει προστασία των επιβατών και σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Ε, θα κάνω μια εξαίρεση και θα μιλήσει και ο κύριος Πάτσκα. legislatívy pre dopravu. Σας ευχαριστώ. Ε, η νομοθεσία αυτή επεκτείνεται κάτι το οποίο θα είναι καλό για τις ε, μεταφορές. Δεν είναι δυνατόν να δούμε με τρόπο τομεακό γιατί βεβαίως τα διάφορα μέσα μεταφοράς συνδέονται και έτσι πρέπει να το δούμε. Το δούμε από τη σκοπιά του χρήστη, του επιβάτη. Εάν δεν λειτουργήσει ένα μέσο μεταφοράς Μπορεί να συμβεί αυτό. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα άλλο μέσο μεταφοράς ο επιβάτης. Και βεβαίως οι εταιρείε θα πρέπει να είναι υπεύθυνε για να φτάσει ο επιβάτης από το σημείο Α στο σημείο Β. Σύμφωνα βεβαίως με τους κανόνες. Εάν δεν είναι σε θέση να το κάνουν, πρέπει να πληρώσουν αποζημίωση. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρωθεί η διαδικασία και έτσι. Θα ακούσουμε ακόμη μια φορά λοιπόν τον Επίτροπο, τον κύριο Πίμπαλξ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζωος και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών για την δουλειά τους στα δικαιώματα των επιβατών. Ακούσαμε μια επικοδομητική συζήτηση από την Κομισιόν παρουσίασε ένα όραμα για μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς στην ανακοίνωσή μας πέρσι. Θα ήθελα να κάνω τα εξή σχόλια επί της έκθεσης. Η Κομισιόν συμφωνεί με τον στόχο να κωδικοποιηθεί το τωρινό πλαίσιο σε έναν ενιαίο κανονισμό, αλλά μεσοπρόθεσμα. Ο κανονισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα, δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές ε, και στις μεταφορές με λεωφορεία δεν έχει ακόμα τεθεί ενισχύ. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ε, μέσων μεταφοράς και οπωσδήποτε η διαδικασία αυτή θα είναι σταδιακή. Η Κομισιόν Σύμφωνη με την δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού εντύπου παραπώνων σε κάθε μέσο μεταφοράς, κάτι το οποίο υπάρχει ήδη για την αεροπορία. Η Κομισιόν σκοπεύει να αναπτύξει έντυπα για τα άλλα μέσα μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Η Κομισιόν επίσης γνωρίζει τον αντίκτυπο που έχουν οι χρεοκοπίες ε, αεροπορικών εταιριών στους επιβάτες οι χρεοκοπίες Spanair και Malev ε, υπήρξαν αντικείμενο καλής διαχείρισης και χάρη στην παροχή πληροφοριών και ε, την συνεργασία δόθηκαν από άλλες εταιρείες φθηνά εισιτήρια για να επιστρέψουν στο σπίτι τους οι επιβάτες. Οπότε μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση των χρεοκοπιών. Όμως χρειάζονται λύσεις έτσι ώστε οι επιβάτες να μην μένουν αποκλεισμένοι και να λαμβάνουν τα λεφτά τους γρήγορα. Οπότε η Κομισιόν το τέλος του 2012 σκοπεύει να υποβάλει προτάσεις για λύση, όχι οπωσδήποτε νομικής φύσεως, για να φροντίσουμε να υπάρξει η εφαρμογή του στο συντομότερο δυνατόν. Τέλος, το ζήτημα της διαφάνειας των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων αναφέρεται σε πάρα πολλά νομοθετήματα, ειδικά δε στον κανονισμό αεροπορικών υπηρεσιών. Να ενημερώσω τις κυρίες και τους κύριους βουλευτές πως ε, αυτή τη στιγμή επανεξετάζουμε την νομοθεσία για να δούμε εάν επαρκεί για να εκπληρώσει τον στόχο της και ε, μήπως πρέπει να αναθεωρηθεί η Κομισιόν κατόπιν θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα αυτά εν ευθέτω χρόνο η δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των δικαιωμάτων αεροπορικών επιβατών είναι πολύτιμος οδηγός για την Κομισιόν, ειδικά εν ώψη της αναθεώρησης του κανονισμού για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και αυτή η ψηφοφορία αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Φτάσαμε στο τέλος ημερήσιας διάταξη για απόψε. Να σας υπενθυμίσω πως η συνεδρίαση θα επαναληφθεί αύριο 3η 23 Οκτωβρίου και θα ξεκινήσει σε μια ώρα ασυνήθιστη 8.30 η ώρα με 10